Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Κάποιε Κάποιες ανακοινώσεις έχω να κάνω, αλλά πρώτα Θα ήθελα να σας ζητήσω να εγκρίνετε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Ε, στην σχέδιο ημερήσιας διάταξης θα δείτε ότι η ψηφοφορία ε, έχει ανασταλεί για ε, κύριο θέλετε να εξηγήσετε αγαπητοί συνάδελφοι Η κατάσταση για αυτό το φάκελο των τεχνικών ε, περιορισμών, των περιοριστικών διατάξεων έχει ως εξής. Ε, βρισκόμαστε ίσως πολύ κοντά σε μια εύλογη συμφωνία. Έχουμε προβεί σε κάποιους τεχ... τεχνικούς συμβιβασμούς ασφαλείας. Ε, τίθεται το ζήτημα των βαρών και είχαμε σχεδόν καταλήξει σε συμβιβασμό για τα βάρη και τις διαστάσεις και όλες τις λοιπές ε, πτυχές που αφορούν ε, τα φορτηγάδια συνοριακών μεταφορών. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε μάλλον να καταλήξουμε σε τρίπλο συμβιβασμό μέχρι την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ λοιπόν από βάθος καρδίας ε, τους και οι οποίοι ήταν ε, τόσο πρόθυμοι να συνεργαστούν για τους συμβασμούς. Ε, είναι πολύ δύσκολο, πολύ οι δυσκολίες αυτό το φακέλου και πολλά τα συμφέροντα που διακυβεύονται. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για το ε, δέσμευσή τους να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα. Μια τελευταία παρατήρηση. Θεωρώ ότι θα ήταν πιο εύλογο να αναβάλουμε το σύνολο πακέτο του πακέτου για την επόμενη θητεία. Έχω δύο μηνύματα. Ε, σε εκείνη την περίπτωση θα έχουμε άλλον επίτροπο μεταφορών, ο οποίο ίσω να μην είναι τόσο ευνοικό για το άνοιγμα των συνόρων. Αυτό έχουν να πω προτείνουν αναβολή του φακέλου. Και δεν θα είμαι ίσω καν εγώ εισηγητή του φακέλου πλέον, οπότε τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Για ορισμένε αντιπροσωπές λοιπόν που βρίσκονται εδώ και που ενδεχομένω σκέφτονται κάτι τέτοιο, ότι καλό θα ήταν να το αναβάλουμε, θα ήθελα να τους παροτρύνω να το σκεφτούν ε, και να σκεφτούν ότι δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα να καθυστερήσουμε ε, το φάκελο αυτόν. Εδώ δεν ζήτημα διασυνοριακών μεταφόρων, αλλά βελτίωση των συνθήκων εργασίας των ανθρώπων σε αυτό το τομέα. Τίθεται θέμα ασφάλειας για τους οδηγούς των οχημάτων αυτών. Ελπίζουμε λοιπόν με, αυτή, αυτό το συμβεβασμό να καταλήξουμε να αριθμίσουμε το ζήτημα αυτό στην Ολομέλεια του, Ιουλίου, του Απριλίου. Συγγνώμη. Όποιος θα ήθελε να μιλήσει παρακαλώ να είναι σύντομος και ακριβής κύριε Γκρός. Η αναβολή του φακελού συμφωνώ αλλά Θέλω να το συζητήσουμε στην Ολομέλεια και να ψηφίσουμε αν τουλάχιστον δεν περάσει η συζήτηση. Αυτό θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε και ανάλογα να διοργανωθεί και η ψηφοφορία στην Επιτροπή γιατί η επόμενη Πέμπτη ε, το πρωί ενδεχομένω να είναι το πιο ευνοϊκό σημείο χρονικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν χρειάζεται για την Ολομέλεια, να το βάλουμε οπωσδήποτε. να πάει στην ε, ε, ολομέλεια του Μαρτίου ο πρόεδρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, κοιτάμε και έχουμε υπόψη μας ε, το Μάρτιο, αλλά ενδεχομένω και την ολομέλεια του Απριλίου. Αυτό κατάλαβα εγώ, κύριε Γκρό. Well, everything, everything on... Όλα θα εξαρτηθούν ε, από τον Απρίλιο, ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε τελευταία στιγμή, αλλά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο κύριο Συγητή λέει ότι θέλει να ασχοληθεί με το ζήτημα και να το έχει ολοκληρώσει σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο και στο επόμενο. Ακολουθεί η έγκριση των πρακτικών. Συμφωνείτε όλοι με την ημερήσια διάταξη, υποθέτω. Πρακτικά λοιπόν συνεδρία στι 6 17 Δεκεμβρίου και 9η Ιανουαρίου. Είστε ικανοποιημένο. Ευχαριστώ. Ανακοινώσει του Προεδρού όσον αφορά τι αποφάσει που έχουν ληφθεί από του συντονιστέ στις 30 Ιανουαρίου πρώτα απ' όλα ενημέρωση για τη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους και τις τρεις προτάσεις που συνθέτουν τον τεχνικό πυλώνα. Οι συντονιστές θέλουν αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν μαζί. Η κατεξοδότηση πράξης, ε, η σχετική απόφαση είχε αναβληθεί μέχρι σήμερα. αλλά έχουμε λάβει μια επιστολή από τον κύριο Κάλλας που φαίνεται να ελαφρύνει το πρόβλημα. Θα το εξετάσουμε αργότερα. Έχει σημειωθεί επίσης ε, και έχουν ε, ληφθεί επίσης υπόψη τα ενημερωτικά δελτία περί επιτροπολογίας. Χθες έλαβε χώρα η συνεδρία των συντονιστών ε, υπό τον Δομινή όπου η παρουσίαση της Κομισιόν για τους υποψήφιους για την Τέντη ενέκριναν τους συντονιστές τέντη που πρότεινε ο κ. Καλές με επιστολή στις 28 Ιανουαρίου και ζητήθηκε να εκπονηθεί επιστολή που θα αναφέρει την υποστήριξη προς αυτές τις υποψηφιότητε. Θα σας ενδιαφέρει επίσης να μάθετε την εκτίμησή μου προς τον Νίλ Τάνκελσον ο οποίο θα φύγει από τη γραμματεία της Τραν στις 15 Φεβρουαρίου ο Νίλς ε, έχει συνεργαστεί με την Επιτροπή Τραν τα τελευταία πέντε χρόνια για πολλά μικρά αρχεία όπως το TNT, το ΣΕΦ και το πακέτο για τους σιδηροδρόμους και τώρα έχει οριστεί επικεφαλής μονάδας του Τμήματος Πολιτικής Β. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσει να εξυπηρετεί την Επιτροπή. Τραν υπό την νέα του ιδιότητα. Συγχαρητήρια Νίλς, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. ευχαριστούμε για τη συνεργασία σου. Και τέλος, από εμένα έχουμε δύο επισκέπτες ε, με την κυρία Μάισνερ από το Madison, Wisconsin στις Αμερικής. Όσοι παρακολουθείτε τα αμερικανικά σπορ θα τους γνωρίζετε. Καλώς ορίσατε στη συναντήσή μας και ελπίζουμε να απολαύσετε τη διαμονή σας εδώ στις Βρυξέλλες. Ωραία λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα Όλοι είναι ικανοποιημένοι με τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Ωραία. Ακολουθεί η έγκριση της συμφωνίας σχετικά με τις περιοριστικές διατάξεις σχέση με τον θόρυβο στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Λάιχτφριντ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση μου γιατί είμαι εισηγητής για την έκθεση αυτή, αλλά ε, στην ψηφοφορία θα πρέπει να σας ανακοινώσω ότι δυστυχώς έχω ξεχάσει την κάρτα μου για να ψηφίσω. Μάλιστα, να σας ε, πω προσκεκλημένοι από το Madison, Wisconsin, ότι υπό κανονικές συνθήκες είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι. Ε, πάση περιπτώσει, συμβαίνουν και αυτά θα ψηφίσει ξεχωριστά ο κύριος Λάιχτριτ. Ε, Κοίτα και εσείς, εκτός μικροφώνου όμως, το σχόλιο. Μάλιστα, πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Και έτσι λοιπόν, να κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο, μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε κατά πόσον ε, περισσεύουν 15 ε, από το έλκο, συνήθως. Έναρξη ψηφοφορίας, παρακαλώ. Τώρα το ειρωνικό θα ήταν να περισσεύουν ψήφια από τους σοσιαλδημοκράτες, μάλιστα. Πέρας ψηφοφορίας. Εντάξει, όλοι νόμιμοι. Πολύ ωραία. η πρόταση για κανονισμό του Συμβουλίου και του, ε, του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά του θόρυβου στους αερολεμένες τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σχετικέ περιοριστικέ διατάξει. Ο κ. Λάχης δεν είναι εισηγητής. Έναρξη παρακαλώ. Εάν ψήφισατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας, το αποτέλεσμα είναι 25 ψήφοι υπέρ και 5 κατά 4 αποχές, 5 κατά 5 αποχές. Ε, εγκρίνεται και συγχαρητήρια στον κύριο Λάχτφριντ. So the... Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι είναι οι άντρες δύο. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ έχει το λόγο που είναι και η συγγετρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Με χαρά μου σας παρουσιάζω τις τροπολογίες για τις δύο αυτές νομοθετικές προτάσεις και καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την συνεργασία για το ψηφίσμα το οποίο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία την προηγούμενη Πέμπτη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εν ώψη και των ευρωεκλογών σε ό,τι αφορά ένα τόσο σημαντικό κλάδο του, της ιστορικής ναυσιπλοείας. Να υπάρχει ομοφωνία και από πλευράς της Επιτροπής και από πλευράς της Ολομέλειας και μια σαφής κατεύθυνση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το που θα πρέπει να οδεύσει μετά την ανακοίνωση 2002. Για τις δύο νομοθετικές προτάσεις τώρα. Θα συζητηθούν σε ό,τι αφορά τον, τις ικανότητες του στόλου. Πολύ λίγο αλλάζει η φυστάμενη οδηγία και με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω. Μιλάμε για το αποθηματικό το οποίο 35 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται για αποθηματικό και αυτό το καταβάλει ο ίδιος ο κλάδος. Και αυτό προβλέπεται για οικονομικά δυσχερείς καιρούς. Τώρα, λόγω του περιορισμένου εύρους ε, εφαρμογής, οι πλειοκτήτες δεν μπορούν να δαπανίσουν αυτά τα χρήματα. Αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να το υπογραμμίσουμε εξ αρχής, γιατί κάποιες τροπολογίες επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογή χρήση ε, του αποθεματικού για σημαντικούς κοινωνικούς στόχους, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βρούμε κοινωνικές, ε, κοινωνικά κονδύλια ή για παράδειγμα σαφείς ε, ε, ερευνητικούς σκοπούς, οι οποίοι θα καλύπτονται από τον ορίζοντα 2020. Είναι σημαντικό να τον τονίσουμε αυτό εξ αρχής, γιατί όντως είναι περιορισμένο το ποσό, το χρηματικό. Σε, ό,τι αφορά τις τροπολογίες, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις αν μου επιτρέπετε. Η κυρία Τικάου κατέθεσε τροπολογίες για την έρευνα, για τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος, για την πιο στενή παρακολούθηση της αγοράς. Αυτά είναι όντως πολύ σημαντικά. Ωστόσο, εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε άλλη άλλα κονδύλια, όχι αυτό το συγκεκριμένο ταμείο. Ας κοιτάξουμε λοιπόν, αύριο θα γίνει και συνεδρίαση των ε, σκιωδών, να δούμε πώς αυτό μπορεί να πλαισιωθεί σε, μια τελογική σκέψη για να διευκρινίσουμε από πού προέρχονται τα εκάστοτε κονδύλια. Χαίρομαι ιδιαίτερω που ο κύριος Αρτούχ ε, κατέθεσε και αυτός μια τροπολογία για την ε, πρόταση αυτή μόχλευσης ε, των δαπανών. σε ό,τι αφορά το Connecting Europe Facility κτλ. Κοιτάξτε, εσεί το έχετε βάλει στο διατακτικό σου ένα άρθρο, εγώ το έχω βάλει σε αιτιολογική σκέψη. Εγώ θα ήθελα να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν νομικώ πώ θα έχει να μπει αυτό στο ε, τακτικό σε άρθρο, όπως παρουσιάζεται στην τροπολογία 15 του κυρίου Έρτοκ. Ε, το καταλαβαίνω και μου αρέσει σαν σκέψη, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται. Καλωσορίζω και την τροπολογία 12 για την βελτίωση της ασφάλειας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τη σχετική διατύπωση, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το, μπορούμε να το ξεπεράσουμε, να βρούμε μία και ένα κοινό τόπο. Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές τώρα, η έκθεση έχει ως σκοπό την περαιτέρω εναρμόνεση των διαφορετικών ε, τεχνικών προτύπων και καλύτερη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του CCNR. Ε, Επίση, ο κ. Φαντάλε κατέθεσε μια τροπολογία και για τη ρήτρα αναθεώρηση. Και εγώ είχα κάνει κάποιες προτάσεις. Εσείς αλλάζετε την περίοδο από 4 έτη σε 3 έτη. Λογικό αυτό, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την ε, τροπολογία υπαριθμό 19 της Κριζίνε Μέισνερ. Νομίζω ότι θα είναι καλή η γραμμή αυτή, να την ακολουθήσουμε έτσι. Η κυρία Τικάου προτείνει να γίνει διαβούλευση των εμπλεκομένων φορέων. Και αυτό, λογικό, πάντα σημαντικό. Είναι πολύ και διαφορετικοί αυτοί οι εμπλεκόμενοι φορεί, οι οποίοι θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις όταν πρόκειται για τεχνικά πρότυπα. Και για τον κανονισμό αυτό, ωστόσο, να προσέξουμε, γιατί οι προσθήκες του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ε, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής. Για παράδειγμα, η τροπολογία 12 της κυρίας Ναλόβα έχει να κάνει με ε, τις ε, δαπάνες των ε, ταμείων συνοχής και των άλλων ταμείων. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει πολλά με το πέντε εφαρμογή τη τρέχουσα οδηγία. Τέλο, η κυρία Τικάου κατέθεσε άλλη μια τροπολογία σε ό,τι αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών, προσθέτοντα και την Επιτροπή του Δουναβή. Θα ήθελα εδώ να ζητήσω την ε, κατεύθυνση από πλευρά ε, συμβουλέ από πλευρά τη Επιτροπή σε ό,τι αφορά την αμοιβαία αναγνώριση, σε ό,τι αφορά και την Επιτροπή του Ρήνου μιλάμε μόνο για χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ στην Επιτροπή του Δούναβη δεν, είναι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, άρα έχω κάποιε αμφιβολίε. Επειδή ο αριθμό των τροπολογιών είναι μάλλον περιορισμένο, νομίζω ότι καλό. Θα, θα ήταν δυνατόν να βρούμε μια κοινή θέση, ένα κοινό τόπο σε συνεργασία και με τι άλλε ομάδε εδώ στο Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να ζητήσουμε μετά την ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα να ζητήσουμε εντολή για να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον όγκο του στόλου. σε ό,τι αφορά τη μεταφορική ικανότητα. Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές ε, προδιαγραφές έχω κάποιες αμφιβολίες, αλλά να το κοιτάξουμε και να το διευκρινίσουμε αυτό πριν την ψηφοφορία. Τουλάχιστον όμω για τη μεταφορική ικανότητα θα ήθελα να υπάρχει μια συμφωνία με το Συμβούλιο πριν τι εκλογέ. γιατί αυτό ο τομέα τη ιστορικής ναυσιπλογίας περνάει δύσκολου καιρού. και είναι πραγματικά κρίματα αυτά τα 35 εκατομμύρια που δεν έχουν δαπανηθεί κατά το παρελθόν και θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλκαντράου θα επανέλθει επί του θέματος. Ναι, και εγώ υποθέτω γιατί ήταν παρόν. Thank you. Έτσι πιστεύω ότι θα κάνει ο κύριος Σέρτοκ. Ε, κυρία Μάισνερ, σας ευχαριστώ και πάρα πολύ πρόεδρα. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια την Κορίν. Γιατί έω ε, τώρα ήταν πάρα πολύ ευχάριστη συνεργασία και πρέπει να διευκρινίσουμε ότι συμφωνούμε γέννη σε ό,τι αφορά την νομοθεσία αυτή δεν μπορούμε όλα όσα θέλουμε για την εσωτερική πλοία να τα προτάξουμε στο συγκεκριμένο κείμενο. Γι' αυτό λοιπόν και είχαμε αυτό το ψήφισμα το οποίο ανέφερε η, Ευρωπαϊκή, η ε, Κορίν. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε τον κλάδο να Έχουμε διάφορα έργα τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε. Έχουμε διάφορα κονδύλια και από το Connecting Europe, το ΣΕΦ. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί περαιτέρω η ιστορική πλοία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την τομέα μεταφορών και αυτό το ψήφισμα λοιπόν το τόνισε αυτό γιατί δεν ε, συμπεριλαμβάνονται όλα μέσα σε, αυτή την, ε, σε αυτά τα δύο προτάσει. Εγώ μία προτασία έκανα σε ό,τι αφορά τι τεχνικέ προδιαγραφέ. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που μα πρότεινε από πλευρά ε, τη Κορίν. Στι τεχνικέ προδιαγραφέ, η Κορίν το έδειξε αυτό το θέμα. Έχα ζητήσει κάθε προσαρμογή των παρατημάτων να ισχύει για τρία έτη και μετά να το ελέγχουμε αλλά πραγματικά αυτό έχει επιβεβαιωθεί από την εμπειρία της Επιτροπής του Ρήνου σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, τριετία αυτή η περίοδο δοκιμασίας και σε περίπτωση που όλα αυτά όντως αποδείξουν την αξία τους για τον κλάδο να συνεχίσουν να ισχύουν. Σε ό,τι αφορά το αποθηματικό τώρα, καλό θα ήταν να καταλήξουμε σε μία λύση γιατί δεν είναι δυνατόν σε ένα κλάδο όπου χρειαζόμαστε κονδύλια, 35 εκατομμύρια, τα οποία δεν είναι πολλά συγκριτικά, να μην χρησιμοποιούνται γιατί το απαγορεύουν ουσιαστικά οι όροι πρόσβασης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κορίν. Και προσβλέπω στις ε, συζητήσεις, στις επόμενες συζητήσεις. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Σαρτούκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα και συγγνώμη που βγήκα για λίγο γιατί δεν είχα φέρει τα σωστά χαρτιά μαζί. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την εισηγήτρια και τους κοιόδης, επικοδομητική συνεργασία. Καλή, πολύ καλή συνεργασία, όντως. Και αυτό νομίζω καταδεικνύει ότι μπορούμε να επιδιώξουμε από κοινού ένα κοινό στόχο δεν ήταν πάρα πολλέ τροπολογίε. 22 νομίζω. 12 σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την ε, μεταφορική ικανότητα και 10 για τι τεχνικέ προδιαγραφέ. Θεωρώ ότι αυτό είναι καλή ένδειξη. Είναι μια ένδειξη ότι οι πρωτεύοντες στόχοι είναι κάτι που μας βρίσκουν σύμφωνος σε ό,τι αφορά το αποθεματικό για να εξαλείται το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μα Και κατά δεύτερον είναι σημαντικό στι τεχνικέ προδιαγραφέ να υπάρχουν αυστηρή ε, εμπειρογνωμοσύνη ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρογνωμοσύνη. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε τώρα, εν συντομία, στις 18 και στις 12. σύμφωνο ουσιαστικά με τη θέση της εισηγητριάς Γιούτα Στάινμπρουκ της Επιτροπής Απασχόλησης σε ό,τι αφορά την ε, συνεργασία με την Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμενοποίηση των ε, ε, μέτρων για τους απασχολούμενους στον κλάδο. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, προτάσεις για τα μέτρα για τις ηλικιακές, τα ηλικιακά όρια, τα προσόντα του προσωπικού και την επίσημη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων για την ανάθεση και την εκχώρηση των πόρων. Εδώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια καλή συνεργασία με την Επιτροπή απασχόληση. και συμφωνώ με την άποψη τη συζήτηση ότι η μεγάλη πρόκληση για την ιστορική ναυσιπλοεία είναι να δοθούν τα σωστά οικονομικά κίνητρα. Και σε ό,τι αφορά το TNT και τη σχετική νομοθεσία, θεωρούμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε για την ιστορική ναυσιπλοεία και σε ό,τι αφορά τις ε, δυνατότητες που μας δίνει το Connecting Europe Facility για την βελτίωση της βιωσιμότητας της περιβαλλοντικής και σε ό,τι αφορά τους κινητήρες των πλοίων. Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, δε, μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το πιο λίγο είναι πιο πολύ, ξέρετε, έτσι λέμε στα γερμανικά καλύτερα πιο λίγο παρά πιο πολύ σε ό,τι αφορά τις τεχνικές περιγραφές, θεωρώ ότι αυτό είναι σκόπιμο. Το μερίδιο του λέοντος θα πρέπει να το ε, διαπραγματευτούν και να το επεξεργαστούν οι εμπειρογνώμονες. Δηλαδή, να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα, ένα παλμό και να ζητήσουμε στη συνέχεια ε, τακτική αναθεώρηση και έλεγχο, όπως ζητούν και οι συνάδελφοι, προκειμένου να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και την πρόοδο και στις τροπολογίες λοιπόν νομίζω τις ε, ανέφερα, τις ε, εξέτασα, τις παρουσίασα μάλλον και γενικά νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε και να αποδεχτούμε τις διαφορές που έχουμε που είναι περιορισμένες και πάλι ευχαριστώ την συγκεκριά για την καλή συνεργασία. Ο κύριος Βαντάου από το ΙΣΙΑ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Πρόεδρε, καταρχάς ε, να μιλήσουμε για τα θέματα ε, της ικανότητας της μεταφορικής. Ε, μου έκανε πολύ εντύπωση και με σόκαραν κάποιες τροπολογίες του κυρίου Έρτο και της κυρίας Τικάου. Να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα ταμείο με πολύ περιορισμένους πόρους, 35 εκατομμύρια, δεν είναι και πολλά, λίγα μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά δηλαδή ε, τα πλοία και τα έξοδα επιπλέον. Ε, δεν θα πρέπει, όπως είπε και η συγγήτρια, να επιβαρυνούμε τη διαδικασία περαιτέρω με επιπρόσθετους κανόνες, κανονισμούς, εκστρατείες, διοργανωτικά. Θα πρέπει να μην θέσουμε τόσα πολλά. Θα πρέπει να τα αφήσουμε αυτά στα χέρια του ίδιου του κλάδου, να μην τον επιβαρύνουμε υπερβολικά. Θα ζητήσω λοιπόν από την ομάδα μου να μην υποστηρίξει αυτές τις τροπολογίε. Τώρα, η πρώτη πρόταση για τεχνικές πληρογραφέ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που υποστηρίζει η συγκεκριά την τροπολογία μου ή 21. Γιατί την υποβάλλω. Για διάφορους λόγους. Καταρχάς, επειδή θέλω να αποφύγω μια επανάληψη της κατάστασης την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα. Τι έχουμε μπροστά μας τώρα. Μία πρόταση η οποία κατατέθηκε πάρα πολύ αργά στο τέλος της θετίας του τρέχοντος κοινοβουλίου. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν έχουμε ουσιαστικά το χρόνο να γράψουμε μια καλή γνωμοδότηση, μια πλήρη της θετια Γι' αυτό λοιπόν και τραβήξαμε το χειρόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα για να ζητήσουμε πολιτική συζήτηση. Δεν θέλω να επαναληφθεί αυτή η κατάσταση. Και αυτό γιατί τώρα η Επιτροπή κινείται. Ο κύριος Κάλλα την προηγούμενη εβδομάδα το είπε με σαφήνεια την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια ότι θα υποβάλει προτάσεις σε ό,τι αφορά τον τομέα των... για τις ναϊάδες. Και αν αυτές οι προτάσεις είναι ευρείες και αν περιλαμβάνουν και κονδύλια, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Κάλλας, δεν θα πρέπει τελευταία στιγμή να τα ε, επισπεύσουμε τόσο πολύ αυτά. Ζητώ λοιπόν να μου υποστηρίξετε την τροπολογία 21. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται για την ε, τροπολογία 11 σε ό,τι αφορά τον Ντούναβιτς, κυρία Στικάου, να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα έλεγα ότι ναι, ας εξισώσουμε, ας αναρμονίσουμε στο βαθμό του δυνατού της ε, κανονισμούς του Δούναβη και του Ρήνο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν όμως αυτό. Αν είναι δυνατόν και ελπίζω να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν ή εν πάση περιπτώσει προς τα ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε για να υπάρχει μια τέτοια αναρμόνιση, θα ήθελα να υποστηρίξω αυτή την πρόταση. Ευχαρίστως λοιπόν Πρόεδρε να ακούσω την επεξήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό. Η κυρία Τσικάου. Θέλετε κάτι να μας πείτε για το Δούναβι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, συγχαρώ την κυρία Βόρτμαν Κόλ για την εργασία της και την κατάρτιση αυτών των εγγράφων. Εγώ μέσω τροπολογιών ζήτησα να μην περιοριστεί ο ανταγωνισμός μέσω νέων αιτημάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βόρτμαν Κόλ που υποστηρίζει την τροπολογία αυτή και επίσης μίλησα για μία ε, πιστοποίηση, εσωτερική πιστοποίηση για τα πλοία στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Όταν μιλάμε για την εσωτερική αγορά θα πρέπει να έχουμε τους ίδιους κανόνες και να δεχτούμε την αμοιβαιότητα των πιστοποιητικών ή της πιστοποίησης. Γι' αυτό θα ήθελα να εγκριθεί αυτή η τροπολογία. Σε σχέση με την ικανότητα ναυσιπλοείας, επειδή μας ενδιαφέρει η εσωτερική αγορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και επειδή θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τις εσωτερικές πλωτές οδούς, ζήτησα να γίνει μία ανταλλαγή τεχνογνωσίας στους διάφορους ευρωπαϊκούς λιμένες, κάτι το οποίο θα ήταν ευεργετικό για όλους. και θα ήθελα να κάνω και ορισμένα άλλα σχόλια. Θα ήθελα το πρόγραμμα Ναϊάδες 2 να είναι πιο συγκεκριμένο, να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα, διότι το Ναϊάδες 2 χρησιμοποιεί διάφορες πηγές. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια καλύτερη επικοινωνία μεταξύ Επιτροπής και Ταμείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τέλος, χρειαζόμαστε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μία στρατηγική για τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Θα ήθελα να το ζητήσουμε από την Επιτροπή. Έχει μεγάλη ε, σημασία για την ανάπτυξη των μεταφορών στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη. Περνάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη. Πρέπει να πω ότι αυτή είναι μια από αυτές τις σπάνιες ε, ευκαιρίες, ε, περιπτώσεις μάλλον, όπου η Κομισιόν ε, είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη δουλειά που έχει γίνει στο Κοινοβούλιο. Είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου υπάρχει συνένεση όσον αφορά την αξία των προτάσεων. Μπορεί κανείς να διαπιστώσει το επικοδημητικό έργο όλων μας εδώ. Ουσιαστικά όλοι σκεφτόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση ευχαριστήσω την ε, κυρία Βόρτμαν Κόρεν να το συμπεριλάβει αυτό γραπτά στην έκθεσή της. Ε. Λοιπόν, πέρα από τα αστεία, αυτό που ισχύει είναι ότι έχουμε την αίσθηση όλοι ότι λειτουργούμε προς την ίδια κατεύθυνση και εκτιμάμε ιδιαίτερα το έργο όλων. Πρώτα απ' όλα φυσικά της ε, αλλά και όλων των μελών που προσπάθησαν να προσθέσουν αξία και στις δύο προτάσεις μας. Να πω δύο λόγια για τον ΑΙΑΔΕΣ 2. Και ειδικότερα για να απαντήσω στο σχόλιο της κυρίας Τικάου. Το πρόγραμμα ΝΑΙΑΔΕΣ 2 αποτελεί μια στρατηγική εστιασμένη στην ενίσχυση των πλεονεκτημάτων των εσωτερικών πλωτών οδών και στην μείωση των προβλημάτων που παρουσιάζουν. Σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα ΝΑΙΑΔΕΣ, εστιάσαμε τις προσπαθίες μας σε μικρότερο αριθμό κλάδων, ώστε να επιτύχουμε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κατά συνέπεια προτείναμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα για πολύ συγκεκριμένους τομείς όπως ε, τις τεχνικές οδηγίες, την κατάρτιση και την εξειδίκευση που θα δείτε στην επόμενη θητεία, εναθεώρηση των υπηρεσιών πληροφοριών ποταμών ώστε να προετοιμάσουμε τις πλωτές οδούς ε, για τα logistics της επόμενης γενιάς το πληρώματα Όλοι λοιπόν οι τομείς έχουν εξεταστεί και ειδικότερα κάναμε ιδιαίτερε προσπάθειες για τη χρηματοδότηση των υποδομών. η χρηματοδότηση αυτή των υποδομών είναι εξαιρετικά σημαντική ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πλωτέ οδοί θα είναι πλωτέ ε, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου υπό ασφαλεί συνθήκε. και γι' αυτό του έχουμε συμπεριλάβει τι πλωτέ οδού ε, στην έννοια του διαδρόμου του corridor. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση θα ήθελα να σκεφτείτε τα όσα έχουμε κάνει με τη χρηματοδότηση ω εξή. Το γεγονό ότι δεν υπάρχει κανένα πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των εσωτερικών πλωτών οδών είναι κατά την άποψή μα πλεονέκτημα. Διότι διαφορετικά θα περιοριζόμασταν σε ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο. Πρέπει να σκεφτείτε ότι εάν εδώ καθόμαστε και συζητούσαμε ποιο κομμάτι του Connecting Europe Facility έπρεπε να πάει στις εσωτερικές πλωτές οδούς, πιστεύετε ότι θα είχαμε καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα όπως αυτό που μπορεί να επιτύχουμε αφήνοντας το θέμα ανοιχτό και φροντίζοντας να χρηματοδοτηθούν όλα τα καλά έργα. Αν είχαμε αρχίσει να κατακαιρματίζουμε το, το Connecting Europe Facility, δεν θα είχαμε καταφέρει όλα αυτά που καταφέραμε. Αποτελεί λοιπόν πλεονέκτημα για τον τομέα αυτή η ύπαρξη των πολύ καλών κριτηρίων για τη χρηματοδότηση του ΝΑΙΑΔΕΣ και το γεγονό ότι δεν περιοριζόμαστε από κάποια ανώτατη τιμή μπορούμε να πάμε και πιο πέρα. Θα εξαρτηθεί από τον κλάδο. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με όλου τα κράτη-μέλη, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουν να προτείνουν καλά έργα προ χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Connecting Europe Facility, τη διευκόλυνση ε, στην Ευρώπη. Τώρα, α περάσουμε στι δύο προτάσει που έχουμε, τη χρηματοδότηση, τον κανονισμό χρηματοδότησης, ε, συγγνώμη, τον κανονισμό περί μεταφορική ικανότητα των πλοίων και τη χρηματοδότηση. Σκοπό μα ήταν να διευκολύνουμε τη διαδικασία καταμερισμού των κονδυλίων αυτών. Μην φανταστείτε ότι μιλάμε για δισεκατομμύρια. Μιλάμε για 35 εκατομμύρια. Εάν αυτά μοιραστούν ε, στο κάθε σκάφο εταιρική ναυσοπλοεία, ε, μερικέ χιλιάδε ε, αντιστοιχούν στο καθένα. Αυτά τα χρήματα είναι μικροποσά ουσιαστικά. Είναι χρηματοδότηση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για προπαρασκευαστικέ δράσει, για υποστήριξη αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δοθεί να δοθούν χίλια ευρώ σε κάθε ιδιοκτήτη σκάφου ε, και να προφυθούν έτσι τα κονδύλια. Δεν είναι αυτό το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται το Ταμείο. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια αυτά θα δαπανηθούν επίσης και στα στοιχεία της επόμενης γενιάς ε, που δεν υπήρχαν όταν συζητούσαμε για τον κανονισμό του 99 Θέλουμε λοιπόν να δαπανηθούν για την καινοτομία, για το greening και για ακόμη περισσότερα κοινωνικά μέτρα. Αυτό είναι το σκεπτικό στο οποίο βασίσαμε την όλη πρόταση. Γι' αυτό το λόγο επιθυμούμε να διατηρήσουμε τη διαδικασία όπως ανέφερε ε, ήδη, ανέφεραν ήδη κάποιοι εδώ. Θέλουμε να διατηρήσουμε λοιπόν τη διαδικασία στο δυνατόν πιο απλή. Η χρηματοδότηση αυτή προέρχεται από τον τομέα και ο τομέας ο ίδιος, ο κλάδος θα είναι αυτός που θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα δαπανηθεί. Δεν μιλάμε εδώ για κοινωνικούς εταίρους. Ο κλάδος ε, συνέβαλε με κονδύλια και πρέπει να μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος πώς θα δαπανηθούν. Όσον αφορά το ζήτημα του συνδυασμού των κονδύλιων αυτών με άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως το Connecting Europe Facility, τη διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη και την Τράπεζα Επενδύσεων. ένας τέτοιο συνδυασμό ε, θα ήταν ευκταίος. Ε, αυτό είναι βέβαιο. Ωστόσο προτιμάμε αυτό να αναφέρεται σε μια θεολογική σκέψη, διότι αυτό μας δίνει την ευκαιρία και το απαραίτητο περιθώριο να προτείνουμε και να μελετήσουμε ποιο θα ήταν ο καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν το συμπεριλάβαμε σε κάποιο άρθρο, αυτό θα έχει ω αποτέλεσμα ότι θα τροποποιούσαμε επίση και τον τρόπο που εσεί και οι συνομοθέτε έχετε αποφασίσει για τι δαπάνε του ε, χρηματοδότηση αυτή από το Ταμείο. Θεωρούμε λοιπόν ότι αφενός ε, θα κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα όλα αυτά και ότι θα επιδράσει αρνητικά ε, στα κείμενα του Connecting Europe Facility που μόλις έχουν εγκριθεί. Πρέπει, μπορείτε να είστε βέβαιοι λοιπόν ότι κατά την απόψή μας και εμείς εγκρίνουμε αυτή την ετουλική σκέψη η ανάγκη μεγιστοποίηση τη μόχλευση αυτού του ταμείου ε, μέσω του συνδυασμού του με, άλλους, ε, με άλλες πηγές ε, είναι ένα πλεονέκτημα και εμείς θα το μελετήσουμε αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην περιπλέξουμε τα πράγματα όσον αφορά τώρα το ζήτημα της αμοιβαίας των τροπολογιών που αναφέρονται στο Δούναβι, την αμοιβαία αναγνώριση δεν προτείνουμε πρώτα απ' όλα εμείς να τροποποιηθεί αυτό το κομμάτι του κειμένου δεν θέλω να σπαταλώ το χρόνο σας τώρα αλλά για ιστορικούς λόγους συμπεριλάβαμε αυτό το άρθρο 4 και τη σχετική αναφορά. Η λόγοι αυτή είναι ότι εκείνη την εποχή ε, βλέπαμε τα αποτελέσματα της σύνδεσης μεταξύ Δούναβη και Είναι λοιπόν μια ιστορική ε, φράση κατά κάποιο τρόπο που δεν έχει και ιδιαίτερη εφαρμογή σήμερα. Όσον αφορά την ε, τεχνική οδηγία αποτελεί μια τροποποίηση που αποσκοπεί να προετοιμάσει τους κανόνες για την κατασκευή σκαφών για την επόμενη γενιά όπου θα υπάρχει ένας κεντρικός οργανισμός στην Ευρώπη που θα θεσπίζει τους κανόνες αυτούς. Τι κάναμε λοιπόν, απλά πήραμε τα διαδικαστικά στοιχεία και τα βγάλαμε από τα παραρτήματα, διότι ήταν αναμεμειγμένα μεταξύ τους, τα βάλαμε στο κυρίως σώμα της οδηγίας, ώστε το τεχνικό κομμάτι να μείνει όσο το δυνατόν πιο απλό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το Κοινοβούλιο το κατανόησε αυτό και οι τροπολογίε κινούνται προ αυτή την κατεύθυνση. Ζητήστε τη γνώμη μα για ένα ζήτημα, την τροπολογία 11. Πρέπει να πω ότι η διατύπωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πιστοποιητικά για το Ρενό και σίγουρα δεν υπάρχουν πιστοποιητικά για το δούναβη. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, κάθε κράτος μέλος εκδίδει ένα πιστοποιητικό το οποίο ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν τίθεται λοιπόν ζήτημα αμοιβαίας αναγνώρισης. Κάθε κράτος μέλος εκδίδει ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος για περαιτέρω διευκρινήσεις. Η άποψή μας λοιπόν για αυτή τη συγκεκριμένη τροπολογία έχει ως εξή. Θεωρούμε ότι θα δώσει λάθος εντυπώσεις για το τι συμβαίνει στο τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και θα ήταν ανακριβές να παραμείνει όσο έχει. Σα διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σα και με την εισηγήτρια για να καταλήξουμε στου καλύτερου συμβιβασμού και στις καλύτερε συμβαστικέ τροπολογίε. Και κάτι τελευταίο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα με την πρόθεση του Κοινοβουλίου να καταλήξει σε έκβαση με αυτό τον κανονισμό για τη μεταφορική ικανότητα των πλέον ε, διότι και στο Συμβούλιο με την Ελληνική Προεδρία θέλουμε επίσης να καταλήξουμε και βάσει και τις έκθεσεις της παρούσα Επιτροπής. Ε, θα αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Βόρτμαν Κόλ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, συναδέλφους να συνεισφέρουν καθώς και την Επιτροπή η οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί. Θα συνεργαστούμε επικοδομητικά και θα λάβω υπόψη τις προειδοποιήσεις των κυρίων Μάιστεν και Φοντάλεν γιατί πράγματι πρόκειται για περιορισμένα κονδύλια και είμαι πεπισμένη ότι θα βρούμε ε, ένα κοινό έδαφος για να συνεργαστούμε. Ευχαριστούμε Κορίν. Θα ήθελα να σας πω ότι η ψηφοφορία θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου στην Επίτροπη και μάλλον στην Ολομέλεια του Μαρτίου. 20 Φεβρουαρίου, εν πάση περιπτώσει, θα ψηφιστεί εδώ στην Επίτροπη. Δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει ε, τίποτα στα διάφορα. Την 5η ε, 20 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσουμε στις 9, ε, τραγικές αυτές οι πέμπτες, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε θα συνεδριάσουμε. Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου στις 9 κλείνει αυτό το τμήμα της συνεδρίασης, στις 10 θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Ευχαριστώ.